Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Σχεδόν έχουμε συμπληρώσει το ακαδημαϊκό τέταρτο, οπότε ας ξεκινήσουμε. Άλλωστε, Δευτέρα είναι, ε, η έλευση μερικές φορές είναι πιο δύσκολη. Θα έλεγα λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε. Βλέπω έχουν καταφτάσει και κάποιοι επισκέπτες. Εμείς τα δικά μας όμως, ημερήσια διάταξη, σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Οπότε εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Όπως ξέρετε, έχουμε κοινή ακρόαση των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος για τα έγγραφα της Μονσάντο και τη Γλυφοσάτη. Θα λάβει χώρα η δημόσια αυτή ακρόαση την Τετάρτη, 9 το πρωί, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί, στην αίθουσα Γιάν 2Q2. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε ότι αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση λίγο νωρίτερα, στις 2.30 και όχι στις 3 ε, συνήθω, όπως συνήθως γίνεται. Και μάλιστα το πρώτο τμήμα της συνεδρίας θα γίνει και κλεισμένο των θηρών, για να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις της διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ. Ε, έγιναν κάποιες μορφές για έλλειψη διαφάνειας και ανεπαρκή ενημέρωση στις διαπραγματεύσεις με το TTIP. Γι' αυτό κρίναμε σκόπιμο για το Μερκοσούρ να έχουμε πιο τακτική ενημέρωση και γι' αυτό θα έχουμε και κλεισμένο το θυρών συνεδρίαση για την ενημέρωση αύριο από τις 2.30. Διερμηνή έχουμε σε 20 γλώσσες με εξαίρεση τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και ε, κελτικά. Και περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 30 και 31 Αυγούστου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, όσοι ήθιστε θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σημείο 4. Το πρώτο κύριο θέμα, ουσιαστικό ζήτημα τη ημερήσιας διάταξη, η παρούσα κατάσταση και οι μελλοντικέ προοπτικές του τομέα εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτριά μα είναι η κυρία Εράνς Καρσία, την οποία χαιρετίζω θερμότατα. Σήμερα θα γίνει και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φρανσίσκο Μαρσέν Μπόσκε, που είναι ο πρόεδρος της ε, διεπαγγελματικής οργάνωσης ε, ε, αγροδιατροφικής οργάνωσης για τα εγωπρόβατα. Θα ξεκινήσουμε με ανάλυση της κατάστασης και τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα των εγωπροβάτων, που δεν είναι πολύ μεγάλος αλλά είναι σημαντικός Γι' αυτό και αποφασίσαμε να εκπονήσουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, την οποία ανέλαβε η κυρία Εράνς Γκαρσία. Και όπως ξέρετε, ο τομέας εγωπροβάτων δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, ε, χαμηλά εισοδήματα σε επίπεδο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και γενικώ ε, μικρή οικονομική βιωσιμότητα η εξάρτηση από τις άμεσες ενισχύσεις. Απ' τη μία λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για καλύτερη ποιότητα των προϊόντων του κλάδου αυτού, αλλά η παραγωγικότητα είναι σχετικά χαμηλή, εξού και πολλαπλές δραστηριότητες που απαιτούνται για τον κλάδο. Και για να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια επισκόπηση και έναν απολογισμό της κατάστασης. Γι' αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε και έμπειρο γνώμονα, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Πριν όμως δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ράς Γκαρσία, για να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά την παρούσα κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα των εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα το απόγευμα εδώ στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γεωργίας, έτσι ώστε από πρώτο χέρι να μάθουμε από τους εκπροσώπους του τομέα και συγκεκριμένα τον κύριο Μαρθέν ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Μαρθένα θα μοιραστεί μαζί μας τους κυρίους προβληματισμούς του. Αναμφιβολά, ο πιο ευάλωτος τομέας της κτηνοτρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς ε, ο τομέας των εγωπροβάτων. Λόγω ε, της μεγάλης γύρανσης των κτηνοτρόφων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Επίσης, η κτηνοτροφία γενικά υπέφερε από, πολλές, από πολλά προβλήματα υγείας των ε, ζώων που οδήγησαν σε ε, προβλήματα και οικονομικές ε, λήψεις 25 εκατομμυρίων από, τον, από το 80 και μετά. Πρόκειται λοιπόν για μεγάλη πρόκληση αλλά και περιβαλλοντική πρόκληση γιατί πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευάλωτο τομέα ο οποίος εξαρτάται από τις ενισχύσεις ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής και που επίσης διαρκώς αντιμετωπίζει με τις τελευταίες δεκαετίες μια διαρκή μείωση της κατανάλωσης του κρέατος του τομέα αυτού ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σχετίζεται μια αύξηση του τομέα του γαλακτοκομικού. Ε, στην προκειμένη περίπτωση αυτό ισχύει έτσι ώστε να προσαρμοστεί ο τομέας ε, ε, στην εξέλιξη των προτιμήσεων των καταναλωτών. Και πρέπει να σας πω ότι η κατανάλωση στον τομέα ήταν της τάξης, είχε μείωση της τάξης του 40% από 3,6 κατά κεφαλή. Η κατανάλωση πέρασε στο 2,8. Ε, το 40% περίπου της ευρωπαϊκής παραγωγής ε, αφορά τις ε, χώρες εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά λόγω του Brexit ο τομέας θα υποστεί μεγάλο πλήγμα. Όσον αφορά την αυτάρκεια της ευρωπαϊκής παραγωγής, πρέπει να πούμε ότι το επίπεδο της παραγωγής είναι της τάξης του 86% αλλά ε, υφίσταται μεγάλες πιέσεις ο τομέας των εγωπροβάτων από εισαγωγές κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία από τρίτες χώρες λοιπόν από τις οποίες ε, πρέπει να ε, αντιμετωπίσει μεγάλη, μεγάλο ανταγωνισμό κυρίως σε περιόδους όπως είναι ας πούμε η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη οι υποχωρήσεις που έχουν γίνει απέναντι σε τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη δε ότι από το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνουν κυρίως ε, όλες αυτές οι εισαγωγές από τρίτες χώρες. Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις, ε, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από επιθέσεις αρκούδων, λύκων κλπ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα δεν μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά και πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να ασχοληθεί η Επιτροπή μας μέσω αυτής της, έκθεση έκθεσης πρωτοβουλίας με το θέμα. Ε, πρόκειται για ε, τομέα ο οποίος είναι επίκαιρο και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος τα επόμενα χρόνια και επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ μεγαλύτερες. Το 2015 ο Επίτροπος Φόγαν αναφέρθηκε στην ενίσχυση το, του τομέα ε, των ε, εγωπροβάτων και του εγωπροβίου κρέατος. Πιστεύουμε ότι οι συστάσεις ε, του φόρου στο οποίο μίλησε ο Επιτροπός και που δημοσιεύτηκαν το 2016 μπορούν να αποτελέσουν ένα μπούσουλα για το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι οι οποίοι αφιερώνονται εις ε, σε εκστρατείες ε, ε, για την αύξηση της κατανάλωσης του κρέατος αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επιτροποχό Γαναλάκη να ευχαριστήσω και για τις διάφορες εκστρατείες στην εσωτερική αγορά που ασχολούνται ακριβώς ε, με ε, την ε, ιδέα να προσελκυθούν ας πούμε οι πιο νέοι καταναλωτές, μια και οι καταναλωτές είναι όλο και γυρεότεροι. Επίσης πάρα πολύ καλή ιδέα είναι μια ιδιαίτερη βοήθεια για τις πιο ευάλωτες περιοχές, βοήθεια η οποία οπωσδήποτε θα έρθει να συμπληρώσει τις βοήθειες οι οποίες ενδεχομένως και τις ενισχύσεις τις οποίες λαμβάνουν οι περιφέρειες λεπτομέρειες ε, αυτές ε, ως ιδιαίτερα ε, τρωτές. Επίσης και η διατροφική αλυσίδα θα πρέπει να είναι σημαντικός στόχος έτσι ώστε στον τομέα των εγωπροβίων να, το εγωπροβάτων να ληφθούν υπόψη οι οργανώσει των παραγωγών και της αγοράς. Για τους νέους γεωργούς ή προκειμένου για τους νέους κτηνοτρόφους θα πρέπει να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου που θα ενισχύσουν το σύστημα των ε, άμεσων ενισχύσεων και άμεσων πληρωμών. Ε, ε, είναι πολλά τα μέτρα τα οποία μπορούν και πρόκειται να αναφερθούν στην έκθεση, αλλά εδώ θα ήθελα να σταματήσω έτσι ώστε να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τα σχόλια του εκπροσώπου του κλάδου, έτσι ώστε να κάνει μια εισαγωγή για αυτά τα οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Έρανς Γκαρσία. Ήταν ε, αρκετά διεξοδική εισαγωγή που μας κάνατε. Αγγίξατε μια σειρά θεμάτων, ένα ευρύ φάσμα που φαντάζομαι θα απασχολήσουν και τον καλεσμένο μας. Έχουμε στην αίθουσα και καλεσμένους κυρία Μίλλερ, επισκέπτες από τη Βαβαρία που παρακολουθούν τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Γεωργίας. Σας καλωσορίζω θερμά τους επισκέπτες της κυρίας Μίλλερ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και θα παρακολουθήσετε τις εργασίες μας. Ο εκπρόσωπος ε, της InterOvic, της Διαπαγγελματικής Αγροδιατροφικής Οργάνωσης για τα εγωπρόβατα. Καλησπέρα σας. Ε, ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την κατάσταση στον κλάδο και ευχαριστώ ιδιαίτερα και την κυρία Ράς Γκαρσία που πρωτοστάτησε στην διοργάνωση αυτή και στην πρόσκληση. Όπως είπατε, είμαι πρόεδρος σε Interovic που είναι διεπαγγελματική αγροδιατροφική οργάνωση με τους περισσότερους εκπροσώπους της αλυσίδας του κλάδου από την παραγωγή, τη μεταποίηση και ούτω καθεξής. Και μάλιστα είμαι παραγωγός κτηνοτρόφος εδώ και 40 περίπου χρόνια και εδώ και 37 χρόνια έχω ένα συνεταιρισμό με 16 κτηνοτρόφους. Ξεκινήσαμε, τώρα είμαστε 600 περίπου σε μια πολύ άγωνη και στεγνή περιοχή όπως είναι η Αραγών στην Ισπανία. Το Δεκέμβριο του 2015 και αρχές του 2016 παρακολούθησα το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Εγωπροβάτων ε, που εγγενίασε ο Επίτροπος Χόγκαν με εκπροσώπους ε, όλους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέμα την σοβαρή κρίση που διανύει ο τομέας αγροπραβάτων, όπως έχει ε, φανεί, γιατί χάσαμε 25 εκατομμύρια κεφάλαια τα τελευταία 30 χρόνια, 25% δηλαδή του κεφαλαίου, 2% ετησίως. Και μάλιστα αυτή η μείωση των κεφαλιών του ζωικού κεφαλαίου ήταν ιδιαίτερα ε, δεινή στην Ισπανία. Εκεί τα πρόβατα ε, πέρασαν ε, σε 8.700.000 από 10 εκατομμύρια, από 12 μάλλον εκατομμύρια. Και αυτό οφείλεται μέρη στην έλλειψη κερδοφορίας αλλά και στην ε, έλλειψη ενισχύσεων. Και μάλιστα σε άγωνες περιοχές και ξηρές περιοχές όπως είναι η Αραγών είχαμε απώλεια 50% του ζωικού κεφαλαίου. Και στην Ανδαλουσία την Εστρεμαδούρα είχαμε αντίστοιχες απώλειες ζωικού κεφαλαίου προβάτων. Η κατάσταση αυτή δεν φαίνεται και πολύ λογική μάλιστα. Σε μία ε, κατάσταση που στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αυτάρκεια εγωπροβάτων. Μάλιστα 212.000 τόνους ε, ετησίως ε, εισάγουμε, άρα εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές και 25% αυτών προέρχονται από τη Νέα Ζηλανδία. Κάτι που επηρεάζει τις τιμές εγωπρόβιου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια η η εισαγωγή νοπών προϊόντων χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες με, αποτέλεσμα να έχουμε ανταγωνισμό με την δική μας παραγωγή που κορυφώνεται σε, στην περίοδο του Πάσχα. Ε, και μάλιστα είναι εποχιακή κυρίως αυτή η παραγωγή. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, εξάγει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 85.000 τόνους. Οπότε μετά τον Brexit θα πρέπει να γίνει μια αναδιαπραγμάτευση ε, και αναθεώρηση της κατάστασης. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε αμία τις ποσοστώσεις ενώ θα έχουμε χάσει τις ποσότητες ε, εισαγωγής ε, εγωπροβάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί αρχικά είχε φανεί ότι θα πάγωνε η ε, παραγωγή, αλλά εξαιτία του άμεσου ανταγωνισμού στον τομέα του νοποκρέατο είχαμε διαφορετική κατάσταση. Παραλαμβάνω, 60.000 τόνοι είναι η εξαγωγή, το 50% αφορά νοπά κρέατα, κυρίως προς την Αφρική, που είναι μια ε, νέα αγορά που αρχίζει και αναπτύσσεται και φαίνεται ότι όλο και περισσότερες περιοχές του κόσμου εκτιμούν την ποιότητα και την ε, επιστηστική ασφάλεια που προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, το ποια είναι τα βασικά προβλήματα του κλάδου, κυρίω η έλλειψη κερδοφορία. Δεν είναι προσοδοφόρε οι κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσει και η χαμηλή παραγωγικότητα συνδυάζεται με χαμηλέ τιμέ που είναι κάτω του κόστου παραγωγή. Και μάλιστα όταν έγινε η σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή εγωπρόβιου κρέατος, και η ενίσχυση πηγαίνει στη γη, είναι σαφώς ότι όταν μία δραστηριότητα δεν είναι προσοδοφόρος, ε, θυσιάζουμε τον λιγότερο προσοδοφόρο κλάδο που είναι ο κλάδος εγωπροβάτων και είτε καταργούμε την παραγωγή είτε περνάμε σε άλλη παραγωγή. Και μάλιστα αυτή η σύνδεση της ενίσχυσης με τις εκτάσεις ε, έπληξε ιδιαίτερο στον τομέα εγωπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η εστίαση των ενισχύσεων. Σε μερικές χώρες θεσπίστηκαν αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή. Αλλά σε τελική ανάλυση κάθε κυβέρνηση ε, κατανέμει το πακέτο στους διάφορους τομείς και στην περίπτωση των εγωπροβάτων ήταν ανεπαρκή τα κονδύλια. Έτσι, η λίγη ενίσχυση που λαμβάνουμε δεν δίνει κίνητρα ε, για εξυγχρονισμό, σε αντίθεση με τη Γαλλία που έδωσε κίνητρα για τους νέους παραγωγούς που επικεντρώθηκαν είτε στην οικολογική εστίαση είτε στην ποιότητα και κυρίως ε, σε περιοχές που είχαν ε, μεγαλύτερα μειονεκτήματα περιβαλλοντικά. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως ας πούμε ότι έχουν αποκλειστεί από τις άμεσες ενισχύσεις ε, τα φωσκοτόπια, φωσκοτόπια ε, λοιπόν λιμόνες ε, λόγω υπερβολικής παρουσίασης, υπερβολικής κλίσης ή λίγο, λόγω υπερβολικής παρουσίας δέντρων ή πετρόδους εδάφους. Αυτά αποκλείστηκαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιούργησε, προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως σε χώρες ε, της ε, ε, Μεσογείου που ακριβώς έχουν τέτοιου είδους γεωφυσική πραγματικότητα και επομένως λόγω έλλειψης αυτών των ενισχύσεων υπέστησαν μεγάλο πλήγμα οι κτηνοτρόφοι, η παραγωγή αυτή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν, να ληφθούν μέρημνες για το θέμα αυτό. Επίσης υπάρχει και διασύνδεση με την ε, περιβαλλοντική ε, πολιτική, ε, ας πούμε, για τις περιπτώσεις του πρασινίσματος ή για τις περιπτώσεις του παγώματος των γεών. Όμως εδώ έχουμε ένα 25% και αυτό το 25% είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σεβαστούν οι γεωργοί και επομένως αποφάσισαν να μην δίνουν τα χωράφια τους στους κτηνοτρόφους. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν, ε, ε, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα ε, λόγω ακριβώς και της αιρεσιμότητας και λόγω της γενικότερης γραφειοκρατίας. Είναι πάρα πολλές οι κυρώσεις τις οποίες υφίστανται πάρα πολύ οι έλεγχοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά όλα είναι απαραίτητα αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να περιπλέκεται τόσο πολύ η ζωή των ακτινοτρόφων και επομένως να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. Θα πρέπει οπωσδήποτε οπωσδήποτε ε, να ε, αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά την ταξινόμηση και όσον αφορά και τις ε, κυρώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη ταυτοποίησης, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη να γίνει, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει ταυτοποίηση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και η χνηλασιμότητα ανά παρτίδες κρέατος. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα ε, για τους ε, κτηνοτρόφους ε, είναι το θέμα των ζώων και των θηρευτών. Είχαμε επιθέσεις λύκων Ε, και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπουμε ότι αυτό πλέον έχει πάρει διαστάσεις εφιαλτικές. Η παρουσία τέτοιων αρπακτικών θηρευτών κυρίως σε συγκεκριμένες ε, περιόδους ε, προκαλούν πάρα πολύ μεγάλη ε, ζημία και οι κτηνοτρόφοι ζουν ακριβώς με αυτήν την διαρκή απειλή. Είναι πάρα πολλά τα χωριά, ακόμα και σε περιπτώσεις οικολογικής παραγωγής, πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή λόγω αυτών των κινδύνων. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά την κατανάλωση. Αφενός λοιπόν έχουμε παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ε, κρέατος ε, και ε, γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ελέγχους πάρα πολύ σημαντικούς που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και άλλες περιφέρειες της γης και σίγουρα οπωσδήποτε δεν είναι οι ίδιες, οι ίδιοι έλεγχοι στην Νέα Ζηλανδία και επομένως εδώ ήδη έχουμε ένα ζήτημα καθώς επίσης λέμε ότι έχουμε από την άλλη πλευρά περιφέρειες της Ασίας και της Αφρικής, κυρίως Βόρειας Αφρικής, που αρχίζουν και κατανοούν την, και εκτιμούν ε, την ποιότητα ε, αυτού του ε, κρέατος και επομένως το εντάσσουν στη διατροφή τους. Το, ένα σημαντικό σημείο είναι για τον τομέα των εγωπροβάτων είναι ο πάρα πολύ ψηλός βαθμός αλληλοσύνδεσης που έχουμε με το περιβάλλον και με τον χώρο της και τον κόσμο κόσμο της 25% ε, της, ε, ε, του τομέα εκπροσωπείται από μια οργάνωση η οποία αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος πραγματικά είναι συνδεδεμένος με τη γη και ε, πρέπει να πω ότι ε, αυτή η διασύνδεση με την ε, βιωσιμότητα και με το περιβάλλον είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνδεδεμένη πλέον ενίσχυση σε ευρύτερες ζώνες οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλες κυρώσεις λόγω της ΚΑΠ και λόγω των λιμώνων που ανέφερα προηγουμένως. Θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και ο πολύ σημαντικό ρόλος των επαγγελματικών οργανώσεων, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρηματοδότησε μία, ε, ε, μία μελέτη η, οποία αναφέρει ότι εάν μία συνεταιριστική οργάνωση εκπροσωπεί το μισό και πάνω των παραγωγών, τότε έχει καλό, καλή επίπτωση σε ολόκληρη την περιφέρεια και σε ολόκληρη την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ε, υπάρξει και ε, διασύνδεση με τον πληρωμών γιατί με τον τρόπο αυτό διατηρούμε και τον πληθυσμό της υπαίθρου στην Ήπεθρο και στα χωριά στην Ισπανία. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου υπάρχουν πάρα πολύ μικροί οικισμοί, πάρα πολύ μικρά χωριά που στην ουσία ζουν ακόμα εκεί στην Ήπεθρο ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι κάνουν αυτή την κτηνοτροφική ε, την, ε, αυτή την κτηνοτροφική παραγωγή ε, εγώ προβάτων. Το πρόβλημα επίσης το γενολογικό, το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάνω από 60 χρονών είναι ο μέσος όρος των κτηνοτρόφων που ασχολούνται με τα ε, εγωπρόβατα ε, και οι νέοι δεν έχουν την τάση να ε, αναλαμβάνουν τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ή να ασχολούνται με τον τομέα αυτό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί και το θέμα της καινοτομία στον τομέα και των ερευνών, της βοήθειας γενικότερα ε, και της παρακολούθησης που πρέπει να έχει ε, ο τομέας αυτός. Είναι γεγονός ότι ε, οι βιοτεχνικές δραστηριότητε έχουν βεβαίως μέλλον, αλλά οι νέοι γεωργοί ξέρουμε ότι είναι στραμμένοι προς τις νέες τεχνολογίες, θέλουν τις νέες τεχνολογίες και οι συνεταιρισμοί θα πρέπει οπωσδήποτε να βοηθούν όσον αφορά την καινοτομία, τη χρήση νέων τεχνολογιών κλπ. Θα πρέπει επομένως να ευνοηθούν ε, και οι επενδύσεις ε, σε τέτοιες ε, περιφέρειες και σε τέτοιες οργανώσεις και συνεταιρισμούς. Επίσης χρειάζεται προώθηση του προϊόντος έτσι ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση. Θα πρέπει να σας πω ότι το 2015 ξεκινήσαμε στην Ισπανία την πρώτη εκστρατεία, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2018 και από μείον 7% στην αρχή της κρίσης το 2008 στο 2015 είχαμε ε, διατήρηση ε, της παραγωγής και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ε, για, το, για τις έρευνες αγοράς το 2015 θα έχουμε μια αύξηση του 1,6% στην γενική κατανάλωση. Μέσω των εκστρατιών αυτών καταφέραμε να βελτιώσουμε την γενικότερη γνώση και την αντίληψη του, του προϊόντος. Μέσω αυτών των των ε, εκστρατιών ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι αλλάζει και ο ίδιος ο ε, τομέας, ο ίδιος ο κλάδος. Δηλαδή ε, σιγά σιγά αλλάζουν οι συνήθειες ε, του ε, καταναλωτή. Μάλιστα μας είπαν ότι 45% των καταναλωτών που είναι πάνω από 50 χρονών καταναλώνουν περισσότερο αρνή γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερο για την υγεία τους και είναι σύμφωνα με τις συνήθειές τους. Ε, λοιπόν, ε, είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί, να εξυγχρονιστεί, ε, να γίνει πιο μοντέρνος ε, ο τομέας. Ε, αυτές οι εκστρατείες στις οποίες αναφέρομαι μπορεί να μην έχουν άμεσο αντίκτυπο, αλλά όλοι οι εμπειρογνώμονες λένε ότι μια εκστρατεία για να δώσει ικανά αποτελέσματα θα πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά τουλάχιστον 9 ετών, έτσι ώστε να έχει έχει καλά αποτελέσματα. Τώρα κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την ε, πρώτη μελέτη και θα ξεκινήσουμε την επόμενη. Επίσης, ε, θέλουμε να βελτιώσουμε ε, τη, ένα, μια σταθερότητα των τιμών. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούν οι παραγωγοί με το μεταπητικό κλάδο για να σταθεροποιηθούν ε, οι τιμέ και να προσφέρουμε μεγαλύτερες δυνατότητες στους καταναλωτές. Μάλιστα, εγώ συνεργάζομαι με την ε, ομάδα, με την οργάνωση Παστόρες και 5 εκατομμύρια κιλά κρέατος ε, και 80% σε τεμαχισμένα, τεμαχισμένα προϊόντα και μάλιστα κάνοντας πιο μικρά τα τεμάχια ε, αυξήθηκε η κατανάλωση γιατί μειώθηκαν οι τιμές των, επιμέ... επιμέρους ε, προϊόντων και άρα αυξήθηκε και η παραγωγή χάρη στην ύπαρξη πιο ευνοϊκών τεμαχίων για τις ανάγκες του καταναλωτή. Επίσης υπάρχουν κάποια ε, υγειονομικά εμπόδια που θα πρέπει να υπερκεραστούν. Είναι, πρόκειται για έναν παραδοσιακό κλάδο με κέρια σημασία στην τροφική αλυσίδα Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κόσμο και τη ε, αλλαγή στον τεμαχισμό αλλά και τι νέε τεχνολογίε και να βελτιώσουμε την ε, παραγωγικότητα και την, ε, το βιωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων. Στο δικό μου συνεταιρισμό έχουμε πάνω από χίλιου παραγωγούς. Οι, 300 έχουν θεσπίσει ένα σχέδιο εξέλιξης και έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 9 ευρώ στο περιθώριο για κάθε πρόβατο και μάλιστα ε, άλλοι που είχαν πολύ πιο εξελιγμένα σχέδια αυξήθηκαν κατά 19 ευρώ στο περιθώριο και άλλοι έφτασαν μέχρι 27, ανάλογα με το πόσο εκλεπτισμένα είναι τα σχέδια, τα αναπτυξιακά που συντάσσουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για να βελτιωθεί και το βιωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων εστιάζοντας καλύτερα τις ενισχύσεις στους στόχους αυτούς. Και φυσικά η υγεία, η υγειονομική κατάσταση έχει κέρια σημασία και θα πρέπει να καταπολεμούμε με τα μέτρα αυτά και τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί αρχίζουμε και έχουμε νέες ασθένειες όπως την μέραν γλώσσα, κάποια ζυζάνια και μάλλον κάποια έντομα όπως ένα κουνούπι από την Αφρική και άλλα έντομα που εξαιτία τη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό η χρήση των προηγμένων τεχνολογιών είναι σημαντική για να βρούμε λύση σε όλε αυτέ τι νέε προκλήσει. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να πω ότι σε συνεργασία με τι δημόσιε διοικήσει, με τον, οργανωμένο κλάδο, με τι διαπαγγελματικέ οργανώσει και του συνεταιρισμού, μπορούμε, τι προσπάθειές μα να εξέλθουμε από την κρίση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Μπόσκε. επειδή όμως ξεκινήσαμε με καθυστέρηση, μετά υπερεύει από το χρόνο του και ο καλεσμένος μας. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Περνάμε αμέσω λοιπόν στη συζήτηση με τους και ηγητές πρώτα και κυρίως ξεκινάμε από τον κύριο Αντριέ που έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ερένς Γκαρθία για αυτήν την έκθεση την οποία με ανυπομονησία θα περιμένουμε ε, και επίσης να ευχαριστήσουμε και τον ε, ε, εκπρόσωπο του τομέα ο οποίος ε, μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή περιγραφή. Ε, όπως υπόθηκε πρέπει να επαγρυπνούμε γιατί πρόκειται για μια κτηνοτροφία η οποία είναι δύσκολη και η οποία βρίσκεται, εκτελείται εν πάση περιπτώσει σε ορεινές περιοχές, δύσκολες, δύσβατες περιοχές. Είναι επομένως πολύ σημαντικός ο κλάδος αυτός ο όπω είπε και η κυρία Ερένς Γκαρθία προηγουμένω που αντιμετωπίζει και μάλιστα μεγάλες δυσκολίες. Ε, το θέμα της διαφάνειας ε, του περιοθυρίου των τιμών, ε, αυτό είναι ένα θέμα επί του οποίου θα πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει λίγο και μέσω της έκθεσης πρωτοβουλίας να επαναπροωθήσουμε σε άλλη κατεύθυνση τις μελλοντικέ εργασίε τη Κομισιόν. Αυτό δεν είναι αμεληταίο, πρέπει να το προσέξουμε. Ένα άλλο, η αποσύνδεση της ενίσχυσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε ε, υπόψη μας όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία αναφέρεται δηλαδή ε, να διατηρηθεί η ε, σύνδεση της βοήθειας στον τομέα αυτό, γιατί είδαμε ότι και στην κτηνοτροφία και στα στον εγωπρόβιο τομέα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αν και κατά πόσο και με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο, να βοηθήσουμε τους εκπροσώπους. Είπαμε για, για τα εγωπρόβατα είπαμε ότι έχουμε τον τομέα της, ε, του γάλακτος, έχουμε και τον τομέα του κρέατος, αλλά βεβαίως εδώ ε, έχουμε ε, ένα ιδιαίτερο τομέα. Πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη στρατηγική, όχι τη γενική στρατηγική για το γάλα ή γενική στρατηγική για το κρέας. Το τελευταίο θέμα, το θέμα των αρπακτικών θηρευτών, νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ελάσσονο σημασία το, το θέμα αυτό για την ανάπτυξη ε, του κλάδου ε, συμβαίνει στη Γαλλία, ε, στη χώρα σας όπως είπατε, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να αναφέρουμε το θέμα αυτό και ξέρω ότι η κυρία Ερένς Γαρσία το γνωρίζει το θέμα, έχει ευαισθησία όσον αφορά το θέμα αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα το αναφέρει. Υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες ακριβώς λόγω ε, των ε, θηρευτών. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, καθόλου ελάσσονο σημασία ε, για την διατήρηση του κλάδου. Και τέλος και για το Brexit, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Οπωσδήποτε πρέπει να αναφερθεί ο τομέας αυτός γιατί είναι πολύ ευαίσθητος στις, για τις σχέσεις μας με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ. Δέκα δευτερόλεπτα πριν το πέρας του χρόνου που δικαιούστε θα σηκώνω το εργαλείο μου. Και παρακαλώ, έχετε μπροστά σας και το χρονόμετρο. Βλέπετε πόσος χρόνος έχει περάσει, παρακαλώ μην το ξεπερνάτε. Δύο λεπτά η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία άλλη ιστορία θέλω να σας πω εγώ. Ως τώρα άκουσα πολλές ιστορίες για τα, την ανάπτυξη, την πιο πολύ υποστήριξη, πιο πολλά ζώα. Εγώ δεν είμαι υπέρ ε, αυτού. Να σας πω τις συνέπειες που υπάρχουν για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Να ξεκινήσω με τα ζώα. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε μια, ε, ένα ξέσπασμα μια τεράστια και πάρα πολύ επιθετική ασθένεια ε, στα εγωπρόβατα, στην οποία κόστησε και τη ζωή σε, 74 άτομα, 100 άτομα μολύνθηκαν και ε, ακόμα 800 άτομα πλήττονται από τις επιπτώσεις της ασθένειας αυτής που είναι μακροχρόνια. Πολλές ζωές καταστράφηκα γιατί τα οικονομικά συμφέροντα των ε, ιδιοκτητών εγωπρεβάτων θεωρήθηκαν πιο σημαντικά από τη δημόσια υγεία. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και ε, μια έρευνα στην Ολλανδία κατέδειξε ότι οι ιδιοκτήτες ε, εγωπρεβάτων, και εδώ μιλάμε για, όχι για μια-δυο κατσίκες, αλλά για χιλιάδες ζώα, αποτελούν πρόβλημα. Και γι' αυτό λοιπόν στη χώρα μας στην Ολλανδία ε, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εκτροφίων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να δοθεί λιγότερη υποστήριξη στις επιχειρήσεις αυτές, εκτός και αν μιλάμε για εξυγίανση. Να προσέξουμε λοιπόν το πώς ε, συνδέεται και με θέματα δημόσιας υγείας. Και τέλος, ε, το καλοκαίρι είδαμε φρικτές ε, εικόνε, από ένα εκτροφείο στην Ολλανδία. Έχουμε όλο και πιο μεγάλη ζήτηση για γάλα γίδας, και γάλα στην Ολλανδία και γι' αυτό λοιπόν ε, τα μικρά τα παίρνουν από τις ε, μητέρες τους πάρα πολύ νωρίς και θα θέλω να τονίσω ότι τα ζώα δεν είναι προϊόντα. Δεν εδώ. Ο κύριος Βοβέ που επίσης είναι και ηγητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που αποφασίσαμε να εκπονήσουμε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι επίκαιρη αυτή τη στιγμή, γιατί σε πολλές χώρες ε, η παραγωγή εγωπρόβιου κρέατος ε, παίζει κεντρικό ρόλο στην οικονομία, όπως στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία. Ε, η παραγωγή εγωπρόβιου κρέατος ανήκει στις βασικές εκτινοτροφικές δραστηριότητες. Οπότε είναι σημαντικό και να μιλήσουμε για το τομέα κρεατοπαραγωγή, αλλά και για το τομέα γάλακτοπαραγωγή. Γιατί σε πολλές χώρες είναι αλληλένδετε οι δύο παραγωγές και καλό θα ήταν να θετήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση και των δύο γαλακτοπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή ταυτόχρονα. Και επίση θα πρέπει να προσδιορίσουμε με σαφήνεια τη λογική της παραγωγής και της προάσπισης ε, των ε, ονομασιών προέλευσης ε, στα προϊόντα του κλάδου. Υπάρχει η μάστιγα των θηρευτών, επιθέσεις των θηρευτών και νομίζω ότι θα πρέπει να εγκύψουμε στο θέμα αυτό, όχι γενικά και όριστα, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Θα πρέπει να να δούμε ποιο είδος υλίκου επιτίθεται, γιατί έχουμε όλο και περισσότερα υβρίδια μεταξύ των θηρευτών. Θα πρέπει να καθορίσουμε τον τύπο του υλίκου θηρευτή. Γιατί κάτι θα αλλάξει τελείω, κάτι θα αλλάξει τελείω την προσέγγιση μα ε, ω προ τη σύμβαση τη Βέρνη και θα μπορέσουμε έτσι να εξολοθρεύσουμε τους θηρευτές που απειλούν τα κοπάδια μας. Είδαμε εκθέσεις από την Ιταλία και την Ισπανία και το 40% των λύκων είναι υβρίδια. Και στη Γαλλία έχουμε παρόμοιο θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να εγγύψουμε στο θέμα αυτό ε, με πολύ εμπεριστατωμένο και συγκεκριμένο λεπτομεριακό τρόπο για να υποβάλουμε και προτάσεις στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ στον τομέα αυτό είμαι 37 χρόνια. Όχι τόσα πολλά όσα ο αλλά μία μεγάλη αλλαγή έχω να σημειώσω. Η αύξηση των μουσουλμάνων στην ε, Αγγλία που τους αρέσουν τα πιο ηλικιωμένα ζώα πράγματα Και τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι προντίζουμε καλύτερα τα ζώα αυτά, τα οποία παλιά τα παραμελούσαμε, γιατί είναι πλέον πολύτιμα ως προϊόντα. Πιο πολύτιμα και από την υγεία στην οποία 20% λοιπόν των προβάτων του σχετικού κρέατος καταναλώνεται από τους μουσουλμάνους και μιλάμε και ε, ο πληθυσμός αυτός διπλασιάζεται και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση. Νομίζω ότι η αποσύνδεση ήταν από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν στον τομέα αυτό γιατί παλιά λάμπαναν επιδοτήσει, δεν φρόντιζαν τα εκτροφία τους καλά και αυτό είχε πάρα πολλές επιπτώσεις. Ε, τώρα λοιπόν εστιαζόμαστε πιο πολύ στην αγορά. Είπατε λοιπόν ε, τι θα γίνει και με τον Brexit έχει εμπορικό πλεόνασμα η Μεγάλη Βρετανία. Θα αποτελέσει αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω. Γιατί ακόμα και αν έχουν ε, την φανή ιδέα να βάλουν δασμούς ε, στο κρέας εγώ προβάτων, δεν χρειάζεται να βάλουμε κι εμείς σε τέλη σε άλλα προϊόντα, στα γαλλικά κρασιά και το καθεξής για να γονατίσουμε τις ε, άλλες χώρες. και τι θα γίνει και με τα εγωπρόβατα τα οποία θα περάσουν τα σύνορα, τα χρυσαία σύνορα προς την Ιρλανδία. Και επίσης ε, προβλήματα υπάρχουν με τα άγρια σκυλιά και έχουμε και το φίλο μου που θέλει να φύγουν όλα τα εγωπρόβατα από τα Highlands γιατί θεωρεί ότι θα πρέπει να επανέλθουν στη φυσική τους άγρια κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τους και συγκεκριτές. Οι υπόλοιποι ομιλητές ε, παρακαλώ να μην ξεπεράσουν το 1,5 λεπτό. Λίγο συντομότερα δηλαδή. Θα πρέπει να μιλήσουν από τους προλαλήσαντες. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα, θα σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε την κατάσταση ε, στον κλάδο. Ε, γνωρίζει και ο κύριος Φέρα είναι χαρακτηριστικό. Ο κύριος ο κτηνοτρόφος αυτός ε, προσπαθεί, έχει σταματήσει την κτηνοτροφική του δραστηριότητα και θέλει να πουλήσει την εκμετάλλευσή του. Και μάλιστα ε, δεν έχει καν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, έχει μειωθεί η δυνατότητα κάλυπτο ακριβώ λόγω της ε, υπερήμερης καταβολής των ενισχύσεων, κάτι που είναι απαράδεκτο. Και οι κύκλοι παραγωγής είναι πολύμηνοι, 12-13 μήνες για τα αρνιά, ενώ η χρηματοδότηση των τραπεζών καλύπτει μόνο μερικές εβδομάδες λειτουργίας. Βλέπετε λοιπόν σε τι κατάσταση περιέρχονται οι, οι κτηνοτρόφοι. Επίσης κάποια σκάνδαλα που γίνονται στα σφάγια στηρίζουν αυτές τις εξαιρετικές κατά της κρατοφαγίας και θεωρούν ότι οι κτηνοτρόφοι αποσταθεροποιούν το κλίμα ενώ ουσιαστικά τα λιβάδια είναι ανθρακοδεσμευτικές εκτάσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή μας ε, συντάξαμε πολύ κριτική έκθεση κατά των εμπορικών αυτών συμφωνιών. Θα πρέπει αντίστοιχα να κάνουν και οι ομολογοί μας. Και μάλιστα η ομάδα μας των Εθνών και των της ελευθερίας θα ταχθεί υπέρ της προάσπισης της ε, γεωργίας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρθέν. Ε, σας γνωρίζω εδώ και κάποια χρόνια τώρα και γνωρίζω ε, και τη, το συνεταιρισμό σας, αλλά γνωρίζω τον, τη σοβαρή εργασία σας στον τομέα αυτό. Και να ευχαριστήσω και την κυρία Εράνθε εκ των προτέρων, γιατί είμαι βεβαία ότι θα είναι σημαντική η έκθεσή της και για τη χώρα μου, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να προσυπογράψω την σημασία της ε, ΚΑΠ των ενισχύσεών της στον τομέα αυτό. Πρέπει να βελτιωθούν κάποια πράγματα και ελπίζω ότι στο Omnibus, ε, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη πολύ καλή δουλειά ε, από τον συνάδελφο ε, Παολο Κάστρο, πιστεύω και ελπίζω ότι θα αναφερθεί και το θέμα αυτό των βοσκοτόπων, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την κτηνοτροφία των εγωπροβάτων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για την κτηνοτροφία των εγωπροβάτων που είναι ιδιαίτερο ωφέλιμη για το περιβάλλον. Είναι ε, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό γιατί η παραγωγή, ε, η πρώτη, πιο σημαντική είναι στην, ε, συγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και η δεύτερη στην Ισπανία. Αλλά τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει και επομένως καταλαβαίνετε ότι παραμένει η δικιά μου χώρα. Και τέλος να πω Πάκο, ε, το, θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους, μεγάλη πρόκληση ε, για τους ε, νέους και νομίζω ότι αν κάνουμε ένα καλό βήμα στον τομέα αυτό θα βοηθήσουμε και τους άλλους παρόμοιους τομείς. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Δυνανό, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά την κυρία Ερνά Γαρσία, η οποία έκανε πολύ κανένα άλυση και με ξεκάθαρο τρόπο την κατάσταση στην Ευρώπη και συμπληρώσατε και το θέμα με την παρουσίαση σε ό,τι αφορά την ε, ανάγκη υποστήριξη της εκτροπής αυτής σε ευαίσθητες περιοχές. Και ιδιαίτερα στις δύσκολες εποχές που ζήνουμε εν ώψη του Brexit, σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή παραγωγή και με την παραγωγή στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία και στον Εμένο Βασίλειο και επειδή πέφτει και η κατανάλωση και πρέπει να υποστηρίξουμε και το κρέας και το γάλα και να απευθύνουμε και έκκληση για πιο προσαρμοσμένες παρεμβάσεις ό,τι αφορά την ε, πολιτική, τη γεωργική και πρέπει να επιμένουμε στον ε, τοπικό χαρακτήρα, τον περιφερειακό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε η κατάργηση των επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των κοπαδιών. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα λοιπόν τα θέματα τα τοπικά τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν σημαντικό, σημαντική πτυχή της όλης εκτροφής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τις πιο ευαίσθητες περιοχές οι οποίες και αυτές αξίζουν να έχουν μια πιο σταθερή παραγωγή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω τρεις προτάσεις συγκεκριμένε να κάνω προς τον εισηγητή μας. Καταρχάς, το πρώτο στοιχείο αφορά ένα κέριο σημείο. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αρρωγοί σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς χείρων και εκτροφής ε, χείρων. Και εγώ προβάτω μετά το 2020. Κατά δεύτερον θα πρέπει στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά τις, ε, αρρωγές να δίνουμε να περάσουμε από το 50% στο 80% σε ό,τι αφορά τις Αίγες. Πέραν τούτου, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αλλάξει η νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση των ε, βοηθειών αυτών, προκειμένου οι εκτροφείς να μπορούν πραγματικά να ωφελούνται από την αρρωγή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα των εγωπροβάτων. Δυστυχώς αυτόν τον τομέα τον έχουμε καταλήψει στη μοίρα του. Είναι φτωχό συγγενής των ε, γεωργικών πολιτικών και είναι πιο δύσκολη διαχείρισή του σε σχέση με την βοοτροφία, για παράδειγμα, την εκτροφή βοηδών, γιατί τα εγωπρόβατα ζουν σε πιο δύσβατες ε, ορεινές περιοχές και άρα η διαχείριση είναι πολύ πιο δύσκολη. Το μείζον πρόβλημα του κλάδου είναι η μεγάλη μείωση των ε, τιμών του αρνήσιου κρέατος. Έχουν καταποντιστεί οι τιμές αρνήσιο κρέατος. Πριν από μερικά χρόνια μπορούσε κανείς να αγοράσει αρνήσιο κρέας για 2,5 ευρώ το κιλό. Σήμερα κοστίζει μόνο 1,5 ευρώ το κιλό. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε νέες διεξόδους για το εγωπρόβιο κρέας μας γιατί δεν είναι τόσο περίπλοκη η παραγωγή, αλλά θα πρέπει να διαθέτουμε τα προϊόντα σε δίκαιες τιμές και να ενθαρρύνουμε τις έρευνες και στον κλάδο αυτό. Γιατί χωρίς έρευνα θα είναι δύσκολο να ορθοποδήσει και να επιβιώσει. Κυρία Μίλλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ε, παρουσιάσει αυτές και για τις επεξηγήσεις που φυσικά επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην Ισπανία και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι και στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλά εσωτόπια τα οποία όντω τα χρησιμοποιούν και διατηρούνται λόγω βιοπικιλότητας από τι αγελάδε, από τα εγωπρόβατα. Και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ε, η αποσύνδεση, να μην παρουσιάζεται μόνο ε, αρνητικά, αλλά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα, να προωθηθεί η έκτροφη των εγωπροβάτων. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κλάδος αυτός και το θέμα του λύκου. Ξέρουμε ότι ο λύκος δεν σκοτώνει, αλλά τρώει, κατασπαράζει. Αυτό από πλευράς προστασία των ζώων είναι κάτι παράδεκτο. Θεωρώ. Και το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι ότι ναι μεν εκφράζουμε τη γνώμη μας, αλλά δεν είμαστε η καθήλη αρμόδια επιτροπή για να αλλάξει αυτή η ρύθμιση. Ελπίζουμε λοιπόν όταν εγκριθεί αυτή η πρόταση να καταφέρουμε να προστατεύσουμε με πιο καλό τρόπο και τους εκτροφείς μας και τα εγωπροβατά μας. Ευχαριστώ κύριο Φλάνναγκαν. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, ε, Φρανσίσκο. Και από ό,τι φαίνεται, είτε στην Ισπανία είτε στην Ιρλανδία, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε πολύ παρόμοια προβλήματα και συχνά γίνεται η συζήτηση για τις κοινέ απειλές. Η κοινή απειλή λοιπόν στο σημείο αυτό εδώ σήμερα είναι ότι η εκτροφή αυτή γίνεται σε μέρη όπου ο κόσμος με τα δυσκολία τα βγάζει πέρα. Οικονομικός πώς υποφέρει και γι' αυτό λοιπόν κάτι θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε και μάλιστα γρήγορα και να φροντίσουμε καλύτερα αυτές τις περιοχές ε, από ό,τι άλλες. Μιλάμε για ανανέωση των γενεών. Ε, μπορούμε να μας λέτε ό,τι θέλετε, αλλά αν δεν υπάρξει κέρδος ε, στο προϊόν που παράγεται ή τέλο πάντων με κάποιο τρόπο μπορεί να τα βγάλει πέρα ο εκτροφέα, αν υπάρχει κάποιο απλοποιημένο σύστημα ενίσχυση, το οποίο δεν έχουμε εμεί στην Ιρλανδία, γιατί το σύστημα μα απέτυχε παταγωδό. Πώ θα ανανεωθούν οι γενιέ, γιατί οι νέε γενιέ θέλουν χρήματα, χρήματα στι τσέπε του. Είναι πολύ απλό. Θα πρέπει λοιπόν με οριστικό τρόπο να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να τους πληρώνουμε τους ανθρώπους αυτούς για να παρέχουν τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες γιατί είναι το πιο βιώσιμο κρέας το οποίο επιτρέπει και την δικοποίηση σε άλλους τομείς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι θύματα σε ό,τι αφορά τα μεγά, τα πολλά, τα, τα, τις μεγάλες επιδοτήσεις και σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, στην Ιρλανδική γλώσσα στην περίπτωση της Ιρλανδίας εξαρτάται από την επιβίωση των περιοχών αυτών, γιατί είναι οι τελευταίοι θύλακες όπου μιλάτε, ε, η γλώσσα αυτή. Για να επιζητήσει μία γλώσσα θα πρέπει να τη μιλούν οι άνθρωποι, γιατί όσα ζώα και να έχουμε δεν πρόκειται να μιλήσουν ποτέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν τον κόσμο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Νταντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν ευχαριστήσω την συγγετρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Άγνιου γιατί μας ε, ε, είπε ε, ότι οπωσδήποτε στα πλαίσια του Brexit θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο το θέμα των ε, ορίων των ε, συνόρων ανάμεσα ε, στην Ιρλανδία και την Μεγάλη Βρετανία. Θα ήθελα επομένω ήδη σήμερα το βράδυ θα μιλήσω με τον κύριο Μπαρνιέ να του επιστήσω την προσοχή του. Το είχαμε πει εμεί ότι είναι ιδιαίτερη αυτή η σειρά των συνόρων. Ευχαριστώ λοιπόν συνάδελφε Αγνίου για τα όσα μας είπατε. Ε, όσον αφορά την έκθεση, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή ακριβώς ε, ε, μπορεί να θέσει σωστά τα προβλήματα αυτών των δύο κλάδων. Αναφέρομαι σε δύο κλάδους, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο καλάθι τα, τις έγες και τα πρόβατα. Μιλάμε για δύο κλάδους που εξελίσσονται με τρόπο όχι απόλυτα παράλληλο, γιατί και η κατανάλωση διαφέρει. Ο κύριος παρεμβαίνει εδώ όντως ε, μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία όντως μπορεί να είναι κοινά στους δύο κλάδους ε, αλλά ε, στην ουσία ε, αυτές οι παραγωγές είναι σημαντικές ε, γιατί παράγονται σε ζώνες ιδιαίτερα ευάλωτες οι οποίες δεν θα υφίσταντο εάν δεν υπήρχαν τα εγωπρόβατα. Πρέπει να πω πάντως στη συνάδελφο που μίλησε για το λύκο ότι εκεί που υπάρχουν πολλοί λύκοι σκοτώνουν αυτοί οι λύκοι, δεν δαγκώνουν απλώς και νομίζω ότι είναι ε, ενδιαφέρον να σας πω ότι θα γίνει μία μετακίνηση, ένα ταξίδι στις Άλπεις ακριβώς για να μελετηθεί το θέμα του λύκου. Καλό είναι να στείλουμε κάποιον ε, αντοπρόσωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ως ε, ένα άτομο που ζει σχεδόν πάνω στο Ιρλανδικά σύνορα, η όλη η συζήτηση για τα βουνά και τα σύνορα δεν μου ακούστηκε και πάρα πολύ οικία, αλλά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθεί οποιοδήποτε έλεγχο στα σύνορα για να μην περνούν τα εγωπρόβατα από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι σημαντικό λοιπόν και επιβεβαιώνει αυτό τη θέση ότι θα πρέπει όλη η Ιρλανδία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ψήφισε ο λαός. Σε ό,τι αφορά τώρα τους εκτροφείς των ε, προβάτων, 24% στην Ιρλανδία των Ιρλανδών ε, εκτροφέων ε, τα βγάζουν πέρα οικονομικά μόνο τους ε, και ξέρω ότι η, η Επιτροπή υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά. Οι υπόλοιποι, λοιπόν τι θα κάνουν, θα τα μαζέψουν και θα φύγουν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που είναι λιγότερο βιώσιμοι, αυτοί που βγάζουν το λιγότερο κέρδος, ε, είναι κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που είναι πιο σημαντικοί, γιατί δίνουν στην κοινωνία μια τεράστια υπηρεσία και σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, η οποία είναι θετική προφανώ, είναι θετικό ο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γιατί πραγματικά εξυπηρετούν και καλλιεργούν και φροντίζουν τη γη, αλλά και επειδή από οικονομική άποψη δρούν στις πιο αποκεντρωμένε περιοχέ. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να απευθύνω προ τον κύριο Μπάσκι είναι τι κάνουμε, πώ μπορούμε να κάνουμε για την υπηρεσία αυτή αυτό που κάνουμε για κάθε άλλη υπηρεσία. Να πληρώσουμε. Πώ μπορούμε να προσαρμόσουμε λοιπόν την κοινή αγροτική πολιτική προκειμένου να μπορέσουν να ιδρύσουν το βιό του αυτοί οι άνθρωποι. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ναι, είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση σε ό,τι αφορά την εκτροφή των εγωπροβάτων ε, σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία είναι μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την προστασία τη φύση για να διατηρούνται αυτές οι περιοχές. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε, μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτή η διάταξη. Συμφωνώ με την άποψη των πιο πολλών εμπειρογνωμόνων εδώ ότι η πλήρης αποσύνδεση ήταν ε, κατά πάσα πιθανότητα λάθος και ο τομέας των εγωπροβάτων πληχθεί ιδιαίτερω και σημείωσε επιδείνωση και Αυτές τις επιπτώσεις τις βλέπουμε και σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν κατά πόσο μπορούν να εξαιρεθούν από την αποσύνδεση. Άλλη μια ερώτηση για το θέμα του λύκου. Και προς τους εμπειρογνώμονες ενδεχομένω. Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να το ελέγξουμε το πρόβλημα αυτό με περιβαλλοντικά μέσα. Δεν το πιστεύω, να σα πω την αλήθεια. Αλλά πού θα πρέπει να βάλουμε το όριο για τη ρύθμιση δηλαδή, του πληθυσμού των λύκων, ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί ε, ο κλάδος να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πραγματικά χρήζει της υποστήριξης και της προστασίας μας. Θα ήθελα να θίξω μια σειρά ζητημάτων που δεν αναφέρθηκαν. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Δεν είναι πολλά τα βοσκοτόπια και γι' αυτό το κόστος παραγωγής είναι υψηλό. Επίσης, ο αθέμητος ανταγωνισμός, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, μαστίζουν τον κλάδο. Για να μην μιλήσω για την ε, καθυστέρηση των πληρωμών. Αυτή η περιμερία επηρεάζει τους κτηνοτρόφους που δεν μπορούν να επανεπενδύσουν σε κλάδους που στηρίζουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Ένα άλλο ζήτημα αφορά το, ε, την, τις επιζωτίες, όπως την ε, κιανή γλώσσα, το καταρροϊκό πυρετό, τον αυθόδη πυρετό, και άλλες ε, ζωονόσους. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν, να καταναλώσουμε τέτοια προϊόντα γιατί οι εκμεταλλεύσεις ε, παραγωγής αγοπρόβιου κρέατος βρίσκονται κυρίως σε ορεινέ περιοχές. Θα πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερη προβολή και να διαφημίσουμε καλύτερα τα προϊόντα τους. Ευχαριστώ. Εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αγορητών. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, ο κύριο Χάψ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον ε, την συγκήτρια μάλλον, την κυρία Ραγγαρσία, για την πρωτοβουλία αυτή. Και τον κύριο Φραντσίσκο Μποσκή για τις λεπτομέρειες που μας έδωσε από δική του πλευράς. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά στο φόρουμ για το κρέας ε, προβάτων τα τελευταία δυόμιση χρόνια και θα πρέπει να ομολογήσω ότι στις τέσσερις αυτές ε, συναντήσεις που είχαμε τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ παραγωγικά. Γιατί εντοπίσαμε τα πιο βασικά σημεία επί των οποίων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον κλάδο αυτό. Και όλος ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω το θέμα το marketing, τα ζητήματα marketing την ε, αστική ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία προφανώς ε, συνδέονται ιδιαίτερως και τα θέματα πολλαπλής συμμόρφωσης και φυσικά τις τάσεις στην κατανάλωση. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικοί παραγοντές οι οποίοι θα πρέπει να τους εξετάσουμε. Και είμαι βεβαίως ότι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οι υπηρεσίες προσπάθησαν να βοηθήσουν την όλη διαδικασία αυτή. Να προσθέσω και κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ στη συζήτηση. Η λειτουργία της αγοράς. Η αγορά λειτουργεί επειδή δημιουργήσαμε και τα επωνομαζόμενα dashboards, τα οποία δίνουν μια επισκόπηση της αγοράς σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις των κλάδου. Και σε ό,τι αφορά την ορισμό της προφητικής εκστρατείας που βρίσκεται υπό διαμόρφωση για τα επόμενα χρόνο και είμαστε ιδιαίτερως αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι θα έχουμε ένα ποσό το οποίο θα είναι το αρμόζον για την ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν συναποτελούν ένα πακέτο κοινών στόχων από πλευράς μας και εμείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να προωθήσουμε και εμείς αυτή την επικοδομητική διαδικασία για να προωθήσουμε περαιτέρω το συμφέρον του κλάδου. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ λόγος τώρα στον εμπειρογνώμονά μας για 5 με 7 λεπτά το πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, απόψεις τις οποίες ε, εκφράσατε και που στην μεγάλη τους πλειοψηφία ταυτίζονται ε, με την ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα ενίσχυση ε, για το γενικό καλό το οποίο προκύπτει από την εκτινοτροφία ε, στον τομέα των εγωπροβάτων. Ενισχύσεις λοιπόν οι οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις υφιστάμενες ενισχύσεις οι οποίες υφίστανται στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το μεγάλο πρόβλημα των θηρευτών είναι είναι σημαντικό, το ε, σημειώσατε και εσείς και βεβαίως μελέτες ή διάφορες δραστηριότητες σαν αυτές που αναφέρθηκαν προηγουμένως ε, σε όλα τα φόρα είναι ε, σημαντικές. Υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τη δραστηριότητά τους σε περίεργες, σε δύσκολες περιφέρειες ακριβώς διότι αυτοί οι θηρευτές προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δημιουργούν πρόβλημα και στην βιοπικιλότητα γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υπεραμείνονται της διατήρησης ε, των λύκων ωστόσο δεν λαμβάνουν υπόψη ε, τα προβλήματα τα οποία μπορούν ε, να προκληθούν σε άλλους τομείς. Γνωρίζω ότι μπορεί να είναι προστατευόμενο είδος και ο λύκος αλλά θα πρέπει να προστατευτεί με άλλο τρόπο. Επίσης οργανώσεις των παραγωγών και κοινοπραξίες οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα στους νέους, την επιθυμία στους νέους να συνεχίσουν σε αυτόν τον τομέα, γιατί διαφορετικά ε, πολύ μικρού ορίζοντος είναι το μέλλον ε, που θα έχει ο κλάδος αυτός. Επίσης, ε, αναφέρθηκε το ε, Omnibus προηγουμένως. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θα πρέπει να αναφερθούν όλα τα θέματα αυτά ε, και το θέμα του πρασινίσματος, του greening και το θέμα των ενισχύσεων γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο τομέας. Η προώθηση του κλάδου και των προϊόντων του είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι εκ των ουκάνεφε αν θέλουμε να αλλάξουν οι συνήθειες ε, πρέπει οπωσδήποτε και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είναι κοινό ο παρονομαστής. Ε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει επίσης να υπάρξει καινοτομία, δημιουργία νέων προϊόντων έτσι ώστε να μπορέσουν οι νέοι και κυρίως οι νέοι των αστικών περιοχών να αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο προϊόντα του κλάδου αυτού. Νομίζω ότι πρόκειται ε, για τομέα ιδιαίτερο στρατηγικό για την Ήπεθρο. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα λόγο στην εισηγητριά μα, την κυρία Ράσκαρση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πάλι του συναδέλφου. Ε, σήμερα ε, ακούσαμε μια πολύ καθησυχαστική εικόνα που όμως ταυτόχρονα μας εμπνέει και μας δίνει πολλά κίνητρα για το πώς οι πολιτικές ομάδες τάσσονται απέναντι στο θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή την ε, κτηνοτροφία εγωπροβάτων. Και όχι μόνο για την Ισπανία είναι σημαντικό το θέμα, για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί όλα τα κράτη-μέλη έχουν εγωπρόβατα και σχεδόν όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και την ίδια πραγματικότητα. Γι' αυτό μας ε, διευκολύνει η εκτροφή εγωπροβάτων για να διαφυλάξουμε την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, ε, να διαφυλάξουμε τον πληθυσμό της υπαίθρου και να στηρίξουμε τον αγώνα μας για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους, τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, αυτό που με καθησυχάζει είναι το πόσο καλά γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τομέα, γιατί από το 2015 έχουμε το ειδικό φόρουμ για τα εγωπρόβατα, όπου ακούγεται η φωνή του κλάδου. Ε, η... Χαίρομαι που αναφέρθηκε από τους πράσινους το θέμα των θηρευτών και μας, μας βασανίζει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και σε αυτόνομες κοινότητες όπως Καστίγια Λεών έχουμε τραγωδία. Στην Άβυλα είναι ε, αιματηρή η τραγωδία που βιώνουμε με τους θηρευτές. Φυσικά μας ενδιαφέρει το φυσικό περιβάλλον και στηρίζουμε τη φύση, αλλά θέλουμε να κρατήσουμε και τον ανθρώπινο πληθυσμό. Ε, γιατί πραγματικά επενδύουμε τεράστια κονδύλια στο φυσικό περιβάλλον, αλλά θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν άνθρωποι για να μπορέσουμε την καθημερινή τους δραστηριότητα να στηρίξουν τις περιοχές που εξαρτώνται από τους κλάδους αυτούς. Οπότε κάναμε μια επισκόπηση της κατάστασης και της πραγματικότητας, ακούσαμε τον καλεσμένο μας, τον καλεσμένο μας και τις επόμενες εβδομάδες θα σας υποβάλω το σχέδιο γνωμοδότηση της έκθεσης για να μπορέσετε να το εξετάσετε και να υποβάλλετε τροπολογίες και τον Ιανουάριο ελπίζω η έκθεση που θα προκύψει να μας περιπεί τιμή, να μας καθιστά υπερήφανους και να δώσει ιδέες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον τομέα εγωπροβάτων. Αλλά θέλουμε πραγματικά η ΚΑΠ να εξυπηρετεί το σκοπό της που είναι να κρατήσουμε τον ε, γεωργικό πληθυσμό στην Ήπεθρο με μάλιστα δυνατότητες για μελλοντικές προοπτικές και ανάπτυξη. Ε, να με συμπαθάτε για το σχόλιο που θα κάνω. Καταρχήν, ε, σας συγχαίρω που έχετε καθυσυχαστεί, κυρία Εράς Γκαρσία, αλλά δεν ε, είμαι σίγουρο ότι συμμερίζονται αυτή την ησυχία και την ηρεμία η παραγωγή του κλάδου. Δεν νομίζω ότι έχουν καθυσυχαστεί η παραγωγή μας από την κατάσταση. Και τι γίνεται με τον κλάδο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί από εκεί υφίστανται ανταγωνισμό. Έχουμε διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και από εκεί σίγουρα μόνο η ησυχία δεν προκύπτει για τους παραγωγούς μας. Επίσης, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ιδιαίτερη διατροφική αξία που έχουν αυτά τα προϊόντα. Και φυσικά και το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι σημαντικό. Αλλά πραγματικά τα πρόβατα καθαρίζουν το περιβάλλον, συμβάλλουν στην προστασία του. Και το θέμα της οργάνωσης των παραγωγών. Άρχισε καλύτερη οργάνωση των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και ελπίζω η σύμπνη αυτή που διαπιστώσαμε σήμερα μεταξύ των πολιτικών ομάδων να συνεχιστεί και κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού και των ενισχύσεων που θα εγκρίνουμε για τον κλάδο. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ τον καλεσμένο μας, ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Πραγματικά σημαντικό το θέμα και είναι σημαντικό που προηγείται η συζήτηση αυτή Τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση ή τη νέα μόρφη που θα λάβει η κοινή γεωργική πολιτική. Σας ευχαριστούμε. Κυρίε και κύριοι, 22 με 27 Νοεμβρίου είναι η, είναι η εξέταση της έκθεσης, η προθεσμία για τις τροπολογίες λίγης 27 Νοεμβρίου και η έγκριση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου του 2018. Πέραμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 5, που προβλέπει την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Η συγητή τη γνωμοδότηση, ο συντάκτη γνωμοδότηση είναι ο κύριο Τίμπορ Σάνι, τον οποίο καλωσορίζω εγκαρδιότατα. Αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η κυρία Εκόν. Αλλά οι συντονιστέ μα αποφάσισαν να συντάξουμε και εμεί γνωμοδότηση. Ε, επί της ετήσιας έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού. Θα θυμάστε ότι πέρυσι για το ίδιο θέμα συντάκτης γνωμοδότησης ήταν ο κύριος Νταντάν. Ε, μάλιστα έγινε δεκτή με ενθουσιασμό γνωμοδότηση και αναγνωρίσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία αυτή με τη σύνταξη γνωμοδότησης που φέτος την ανέλαβαν σοσιαλιστές και δύο κύριος Σάνι. Παρακαλώ, κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησης σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συμφωνώ μαζί σας ότι όντως το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλοι μας ε, θυμούνται, θυμόμαστε αρκετά καλά ότι αυτό πολλές φορές συζητήθηκε στην Επιτροπή αυτό, αυτή από το μια και είναι η έκθεση αυτή της ε, πολιτικής ανταγωνισμού, είναι αιτήσια. Και θα συζητήσουμε λοιπόν την κατάσταση αυτό το τελευταίο χρόνο. Ναι, να σας υπενθυμίσω σε όλους ότι πέρσι ο κύριος Νταντά ήταν υπεύθυνε σε ό,τι αφορά την γνωματότηση για την ε, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού για την οποία είναι την Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά σε ό,τι αφορά κιόλα ε, του ε, εμπειρογνώμονε για τα θέματα όπνιμπα, τον κ. Δεκάστρο και άλλου. Τώρα λοιπόν, Πρόεδρε, πιστεύω ότι μια δυναμική πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα ήταν ακρογωνιαίος λίθο του ευρωπαϊκού σχεδίου και το ιδιαίτερο καθεστώ του τομέα της γεωργίας είναι αναντήρητο. Προφανώ η πολιτική ανταγωνισμού είναι απαραίτητη για να λειτουργεί σωστά η ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μα βοηθά να αποφεύγουμε την υπερβολική συγκέντρωση οικονομική και πολιτικής δύναμης και να υπάρχει επικελία και μεγαλύτερη επιλογή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά. Ο τομέας λοιπόν της γεωργίας δεν καλύπτεται επαρκώς στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η ομοιακή προσέγγιση είναι πραγματικά απαραίτητη σε ό,τι αφορά τον τομέα της αγροτικής πολιτικής, η οποία εξασφαλίζει ένα βιωτικό επίπεδο για την ευρωπαϊκή ε, ένωση, γιατί προφανώς ο κλάδος αυτός υπόκειται σε διαρκείς ε, περιβαλλοντικούς και ε, οικονομικούς κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει επιπλέον παράταση των εξαιρέσεων για την κλάβο της Γεωργίας, γιατί η πολιτική του ανταγωνισμού θα πρέπει φυσικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα της αγοράς, αλλά θα πρέπει παράλληλα να προστατεύσει και το συμβητικό επίπεδο που εγγυάται ο κλάδος ε, της γεωργίας. Σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις και τις ενώσεις, είναι σημαντικέ. το ερώτημα του κατά πόσον η ελευθερία για την παραγωγή και την ε, επίτευξη συλλογικών συμβάσεων και διαπραγματεύσεων ε, είναι κάτι το απτό και τα κρατη και τα και οι θεσμοί θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητε σε ό,τι αφορά και την κατάσταση μετά το Brexit, να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με του ε, κανόνε ανταγωνισμού και την κατανόηση και τη ρύθμιση φορολογικών ζητημάτων μεταξύ κρατών μελών. Όπω βλέπετε, λοιπόν, τα θέματα που αναφέρονται στο σημείο αυτό ε, έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνονται διάφορες πτυχές όπως και η σωστή κατεύθυνση του Omnibus ως UTP, η ανάπτυξη της υπέτρου και τα κοινωνικά στοιχεία. Θα πρέπει να σας πω ότι και εγώ με τις τροπολογίες μου προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθώ και αυτό το και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ελπίζω να είναι εξίσου επικοδομητική συνεργασία με τους κοιόδης και θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω όλες τις διαφορετικές προσεγγίσεις ε, γιατί ο απότερος είναι να διευκολυνθεί η ζωή των ατόμων που εργάζονται στον κλάδο γιατί αν διακυβευτεί ο κλάδος αυτός η ζημιά θα είναι υπερβολική και ο κίνδυνος θα είναι ελοχεύει είναι να διτραχθεί η αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων. Και πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι βασικό πεδίο εφαρμογής της άσκησης αυτής είναι να ε, εξερευνήσουμε το νομικό πλαίσιο για να διευκολυνθεί και ο ανταγωνισμός από τη μία στον τομέα της γεωργίας, αλλά παράλληλα να υπάρξουν και διευκολύσεις για τις διάφορες ε, αγροτικές οργανώσεις, επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά και κοινούς θεσμού και συνεταιρισμού. Ε, πρόεδρε, με χαρά να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντάν πρώτα που είναι σκιώδης συζήτης και έχει και πλούσια πείρα γιατί ήταν ο συντάκτης γνωμοδότης για το ίδιο θέμα πέρυσι. Παρακαλώ κύριε Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Σάνι για το πολύ αξιόλογο έργο του που όπως είπε ε, εντάσσεται ε, στην, σε, στην προσπάθεια που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μετά τις εκθέσεις Μαγκίνες, Δελαέ, τη δική μου και ακολουθεί τον ηρμό αυτό των εκθέσεων. Επίσης ε, σχετίζεται άμεσα με τις προτάσεις τον τελών 2016 του κύριου Βέρμαν και της Επιτροπής ε, της οποίας προείδρευε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας. Και μάλιστα το Συμβούλιο είχε χαιρετήσει το έργο του κυρίου Βέρμαν και της Επιτροπής του, είπε ότι θα ήθελε να το εστερνιστεί και αυτό προτείναμε στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus. Ως προς την γνωμοδότηση Σάνη, θα ήθελα να προτείνω στον συντάκτη μας να επεκτείνει κάπως τον προβληματισμό του στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων στο γεωργικό κλάδο. Γιατί πριν από δύο-τρία χρόνια αυξήθηκε, αλλά οι επιτρεπόμενες ενισχύσεις δεν αυξήθηκαν. Οπότε ενώ έχουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, οι κρατικές αυτές ενισχύσεις δεν φτάνουν για να τις καλύψουν. Επίσης, να συνδυάσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό Omnibus με τον προϋπολογισμό, γιατί, με την της έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού, συγγνώμη, γιατί χάρη σε μία ε, στενή συνεργασία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόκειται όσον ούπο να συνάψουμε διοργανική συμφωνία για όλα τα θέματα που αφορούν τις οργανώσεις παραγωγών και το δίκαιο ανταγωνισμό. Και μην ξεχνάμε το άρθρο 42 της συνθήκης που προβλέπει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο γεωρικών προϊόντων μόνο στο μέτρο που προσδιορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεδομένων των στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής που προβλέπονται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να αντιστρέφουμε τα πράγματα, να διαφυλάξουμε το πνεύμα της Συνθήκης και να μην το ξεχνούμε. Επίσης, θα ήθελα να επιθυμίσω στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Γεωργίας, ότι στις προτάσεις που έχουμε ε, υποβάλει, πάνω από τις μισές εμπίπτουν στη διοργανική συμφωνία. Και ε, ανακαλύπτω εμβρόντιτος και σταθμίζω τα λόγια μου ότι κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να παρατείνουν τις προθεσμίες ενώ εδώ και τέσσερις μήνες ε, και έχουμε υποβάλει τις προτάσεις και ε, ακούγονται κάποιες φημολογίες πολύ περίεργες αριστερά και δεξιά προς τις προθέσεις μας και πραγματικά μένω άναδος και συγκλονισμένος από όλα αυτά τα Φαντάζομαι και οι συνάδελφοι το ίδιο, ιδιαίτερα μπροστά στις προσβολές ε, του κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην απόπειρα σφετερισμού των αρμοδιοτήτων του. Αν ε, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοφεύουν μπροστά στα αιτήματα και στη λαϊκή τιμιγορία, θα πρέπει εμεί να ε, διατρανώσουμε τη φωνή των συμπολιτών μας και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να εμείνουμε στη γραμμή που εθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής. Η έκθεση ε, Βέρμαν μάλιστα ε, έτυχε υποστήριξης και από τα θεσμικά όργανα και εμείς ε, θα κρατήσουμε ε, στο διαπραγματευτικό, στη διαπραγματευτική μας ομάδα τη γραμμή που έχουμε μέχρι στιγμής ακολουθήσει. Ευχαριστώ κύριο Φεράμ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να μιλήσουμε για εμπιστοσύνη. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει ενία... Ε, αγορά στις 28 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να κάνουμε μια μακροοικονομική διαπίστωση και να πούμε ότι όλες ε, ε, οι χώρες όπως ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Κίνα κατανόησαν, κατάλαβαν όλοι ότι θα πρέπει να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους για τα γεωργικά. Και μάλιστα ο υποψήφιος Μακρό είχε ζητήσει εκτάκτως 5 για την γαλλική γεωργία. Στην Εθνική Βουλή υπάρχει μια μεικτή επιτροπή ε, και καλό θα ήταν η Επιτροπή Γεωργίας ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προσπαθούσουν να μην γίνονται ταυτόχρονα οι επιτροπές γεωργικού ενδιαφέροντος. Εν πάση περιπτώσει είναι επίγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσμοθετήσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα διασφαλίζει και την ακεραιότητά της αλλά ε, και την ε, γεωργία της. Ε, οι αθέμητες πρακτικές, οι παραχωρήσεις στις εμπορικές συμφωνίες, ΣΕΤΑ, Μερκοσούρ, Αυστραλία, απειλούν τεράστια τμήματα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της ομιλίας μου ότι το να μιλάμε για ενιαία αγορά και ενιαίο ανταγωνισμό ε, είναι πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι απατηλό και εδώ ε, η παγίδα κλείνει, σφίγγει όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ειλικρινώς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο την Πορτσάνη Σιζάνη για την ε, εξαιρετική εργασία του. Έχω τον ε, ε, συνάδελφο Μισελ Νταντέν, ο οποίος πραγματικά συνεχίζει την εργασία και την, τη συνέχεια των εκθέσεων. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε προηγουμένως ο Μισελ Νταντέν. Η εγκεκριμένη ψηφισμένη από μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής ε, έκθεση Omnibus σήμερα ε, έγινε δεκτή με ε, ευρύ τρόπο και από τους Υπουργούς Γεωργίας. Στρέφομαι τώρα στους συναδέλφους της Επιτροπής, κυρίως δε στους ε, συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ανταγωνισμού ε, έτσι ώστε να καταβάλουν προσπάθεια στα πλαίσια μια ισχυρής διοργανικής συμφωνίας που μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη βδομάδα έτσι ώστε να μην ε, υπάρξουν οποιασδήποτε προτάσεις αναπομπής που εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία, έχουμε σύγκληση επί των περισσότερων σημείων ε, που ε, ακριβώς εκπροσωπούν την βούληση του Κοινοβουλίου στην Όμνιμπους. Ε, Ανώφελο να επανέλθουμε κύριε Πρόεδρε ξανά και ξανά σε θέματα τα οποία μας απασχόλησαν τους προηγούμενους μήνες. Το επίπεδο συγκέντρωσης της γεωργίας απαιτεί σημασία, απαιτεί να ακούσουμε ε, και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των γεωργών. Ε, και στον κανονισμό Omnibus αναφέρονται όλα αυτά με ικανοποιητικό τρόπο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε τους γεωργούς ε, σαν ε, ε, οικόπεδα πετρελαϊκά. Χρειάζονται, και στρέφουμε προς την Κομισιόν, χρειάζονται τα εργαλεία αυτά οι γεωργοί. Προτάθηκαν και από την Επιτροπή Βέρμαν, τα συζητήσαμε επί μήνες και επιτύχαμε μία συμφωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ε, η συζήτηση με μια θετική έκβαση ε, έτσι ώστε να έχουμε μια ικανοποιητική γεωργία ικανή ε, να αντιμετωπίζει αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις στην αρχή της διαδικασίας που στραγγαλίζουν τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Τιμπο για την έκθεση αυτή. Εξ ονόματος του σκιώδιου ε, εισηγητού μα ε, μιλώ, του κύριο Χάιτεμα, αλλά πρέπει να το ρωτήσω την απόψή του, γιατί πιστεύω ότι μετά τις ε, εισηγήσεις του Πάολο και του Μισελ, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση ο Omnibus και κατά πόσον θα συμπεριληφθεί, θεωρώ ότι θα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μα έναντι τη επιτροπή ΕΚΟΝ. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ σε ό,τι αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα και σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ πρακτικέ να θέσουμε τα σημεία προτεραιότητά μα. Αυτή λοιπόν, ο κανονισμός Omnibus είναι το ένα σημείο. Παράλληλα θα πρέπει να δουλέψουμε όμω και από την άλλη στο επίπεδο της προβολής των δικών μας επιχειρημάτων από πλευράς της Επιτροπής Γεωργίας. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, την σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω υπόψη μου κάποια μέλη του ΕΛΚ της χώρας μου, που αν διάβαζαν την έκθεση αυτή, θα έλεγαν ότι α, αναφέρεται η ερμόνηση των φόρων και αυτό είναι κάτι που τους τρομοκρατεί προφανώς. Καλά κάνουμε και μιλάμε για ίσους όρους ανταγωνισμού. Και ένα τομέα του ανταγωνισμού, τον οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, το ανέφερα αυτό και σε προηγούμενη συνάντηση με την Επιτροπό Φεστάγκερ. Φαίνεται ότι δείχνουμε μεγάλη προσοχή για να μην παραβιάζουμε τους κανόνες ανταγωνισμού και να μην επηρεάζουμε, να μην στρεβλώνουμε τον ανταγωνισμό και τον καπιταλισμό. Από την άλλη όμως Φαίνεται ότι στην Ιρλανδία και σε πολλές άλλες χώρες δεχόμαστε μια κατάσταση όπου σε ένα κομμάτι γη παίρνει ο ε, εκτροφέας χίλια ευρώ ανά εκτάριο, ενώ ο άλλος από δίπλα μπορεί να μην τίποτα. Όχι επειδή είναι καλός ή κακός ως εκτροφέας, ε, ως παραγωγός, αλλά μόνο και μόνο για ιστορικούς ε, λόγους. Όταν το ανέφερα αυτό και το έθεσα στην κοινή Επίτροπο Φεστάγκερ, για να είμαι ε, δίκαιο, ε, τουλάχιστον ήταν ε, πραγματικά ειλικρινή. Μα είπα ότι δεν ήξερε και πολλά για το θέμα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι ο τομέα αυτό, η περιοχή αυτή, θα πρέπει να το προωθήσουμε αυτό το θέμα και να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Θα συνεχίσουν να ωφελούνται οι μεγάλοι και οι δυνατοί. Και θα είμαστε εμείς πάντα πίσω. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό να επιτρέψουμε να υπάρχει μια κατάσταση όπου ένας ε, παίρνει χίλια ευρώ και άλλο δεν παίρνει τίποτα από δίπλα. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που δεν θα πρέπει να δεχτούμε. Ε, σήμερα είναι πολυμελής η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εκπροσώπους και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Παρακαλώ. Θα ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την κυρία Χένιξ. Πρώτα από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Καλησπέρα σας. Εγγνήσα Χένιξ ονομάζομαι και εκπροσωπώ την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σήμερα. Σας ευχαριστώ καταρχήν θερμά ε, που λάβατε υπόψη την έκθεσή μας και ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Τιμπορσάνη, για τη δική του γνωμοδότηση που είναι ακόμη στη φάση του σχεδίου. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη τα διάφορα σημεία που αναφέρετε και σας διαβεβαιώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θέλουμε οι κανόνες ανταγωνισμού να γίνουν όσο πιο απλή γίνεται και εύχριστοι για τους παραγωγούς, για τους γεωργούς, ώστε να υποφεληθούν από αυτούς και να εξασφαλίσουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο με ε, όρους δίκαιου και θεμητού ανταγωνισμού. Και νομίζω ε, και η Επιτροπή Χόγκαν και Βερστάγκερ στις ακροάσεις τους στην Επιτροπή σας σας παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει και έχουμε στενή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και σε τεχνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό Omnibus, ε, δεν πρόκειται να το σχολιάσω τώρα, γιατί το θέμα της συζήτησης είναι η αιτήσια έκθεση περί ανταγωνισμού. Γι' αυτό και θα βάλω τελεία εδώ. Μάλιστα, δεν θέλει κανείς άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο, οπότε θα ξαναδώσουμε το λόγο στον συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Σάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και την συμμετοχή τους στη συζήτηση. Όπως όλοι γνωρίζουμε είναι φυσικό σε αυτή τη φάση και το τονίζω σε αυτή τη φάση είναι φυσικό να είναι συμπαγής και πολύ σύντομη η γνωμοδότηση. Αλλά μετά τη συζήτηση δεν διαβλέπω ιδιαίτερες διαφορές απόψεων ή αγεφύρωτες σε συμφωνίες μεταξύ μας. Πιστεύω ότι σε επόμενες εβδομάδες θα λιάνουμε όλες τις ενδεχόμενες διαφορές. Πάντως ε, το γενικό αίσθημα ε, νομίζω ότι είναι το ίδιο στην Επιτροπή. Ε, καταρχήν να λάβετε, υπόψη, να λάβετε ότι δεν είναι δική μου προσωπική γνωμοδότηση. Θα είναι γνωμοδότηση Επιτροπής Γεωργίας. Είμαι ο ταπεινός συντάκτης γνωμοδότησης και είμαι διαλλακτικός και ανοιχτός απέναντι στις προτάσεις. Και αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε σύγκρουση ή αντιπαράθεση, ο ρόλος του συντάκτη γνωμοδότηση είναι να καταλήξει σε συντονιστικές ε, συμβαστικές προτάσεις. Καταρχήν, το δίκαιο του ανταγωνισμού περιλαμβάνει κατευθυντήριε γραμμέ για την οργάνωση τη οικονομία και εντό τη οικονομία η διάρουσα θέση κατέχει η γεωργία. Οπότε ο κανονισμό δεν είναι μόνο ε, στεγνοί κανόνε. Α μην ξεχνούμε το σκοπό που εξυπηρετούν και τι ρόλο έχει η γεωργία μέσα στην οικονομία. Επίσης, αληθεύει ότι η Γεωργία δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως ε, τα πλεονεκτήματα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό, τις διατάξεις δηλαδή των συνθήκων και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ε, να αντιληφθούμε ε, και το θέμα του ανταγωνισμού στη Γεωργία που διαφέρει ριζικά από τον ανταγωνισμό στους υπόλοιπους κλάδους. Την τελευταία διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εντοπίσαμε ε, το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση ο ανταγωνισμός δεν θα πρέπει να υπερέχει των κοινωνικών, ε, του γενικού κοινοτικού συμφέροντος. Δεν θα πρέπει να κυριαρχεί ή να δεσπόζει ο ανταγωνισμός ε, ε, στα, στο γενικό κοινωνικό συμφέρον το γενικό συμφέρον της ευρωπαϊκής κοινωνίας και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Σας ευχαριστώ και σας ε, ενθαρρύνω και ψυχώνω να συνεργαστούμε για την διεκπαιρέωση αυτή της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Βλέπω και το γενικό εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άγγελ. Ποιος ζήτησε το λόγο, η κυρία Ράς Γκαρσία. Όχι. Ουδής. Τροπολογία μέχρι ε, τη, τις 16 ε, Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα. Ε, χαιρόμαστε που ολοκληρώσαμε αυτό το θέμα. Να μην ξεχνάτε 16 Οκτωβρίου τροπολογίες, 7 Δεκεμβρίου έγκριση γνωμοδότησης και τον Ιανουάριο η Αρμόδια Επιτροπή. Περνάμε στο σημείο 6, του δημοσιονομικούς κανόνε που ισχύουν για το Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το λεγόμενο κανονισμό Omnibus. Ο εισηγητής Επιτροπή μα είναι ο κύριο Ντέ. Θα μας ενημερώσει για τον τριμερή διάλογο και τις εξελίξεις. Έχουμε και τον επικεφαλής αντιπροσωπείας, τον κύριο αλλά και τον κύριο Ταντέν, την κυρία Μίλλερ. Είναι πλούσια εκπροσώπηση των εκ μέρους των αρμοδίων για το θέμα του Όμνιμους. Θα, δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ντέσπο, από πρώτο χέρι θα μας παρουσιάσει τις πληροφορίες για τις εξελίξεις των συζητήσεων. και το τι μας περιμένει στην, στον επόμενο γύρο διαπραγμάτευσης της Πέμπτης. Κύριε Ντές, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να έλθω και πιο νωρίς στη συνεδρίαση. Να σας αναφέρω το εξή. Η Επιτροπή Γεωργίας ζήτησε και πρότεινε τέσσερις, τέσσερις ε, κανονισμούς ε, απλοποιήσεις και διευκρινήσεις. Έχουν λάβει η χώρα τρεις ε, τριμερείς διάλογοι το Σεπτέμβριο και πάρα πολλές τεχνικές συζητήσεις και συναντήσεις. Ο τελευταίο τριμερείς διάλογος 27 Σεπτεμβρίου ήταν ένας τρεμερής διάλογος στον οποίο η ομάδα μας προέβαλε πολλά τεχνικά ζητήματα και στις 27 Ενάτου το Συμβούλιο δεν είχε λάβει ακόμα εντολή για τα πιο πολλά σημεία. Και στον τρίτο τρεμερή διάλογο λοιπόν 27 Ενάτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τι άμεσε πληρωμέ, έκαναν κάποια βήματα προ τα πίσω, μα έκαναν κάποιε επαναχωρήσει ή εν πάση περιπτώσει τι υπονόησαν για να βρεθούν για παράδειγμα τεχνικές λύσεις, τις τεχνικές ομάδες. Δεν έγιναν ε, όμως εδώ, δεν μας έδωσε καθόλου αέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Συμβουλία σε ό,τι αφορά το greening, σε ό,τι αφορά τα επόμενα διάστημα. Οι προτάσεις ε, για τις οικολογικές και την ε, τις οικολογικές εκτάσεις και τη χρήση σουλφάτης βρήκαν συμφωνία και τον επόμενο τρεμερή διαλόγο θα ίσως θα συζητηθούν περαιτέρω από τα δύο θεσμικά όργανα. Επίσης υπήρξε συμφωνία όλων των θεσμικών οργάνων για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε τέτοια θέματα. Περαιτέρω σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο συνέχισε να υποστηρίζει την στάση του για τα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να ξεπερνούν την κοινοβουλευτική θητεία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αντίσταση εδώ, γιατί υπάρχει φυσικά η επιφύλαξη της χρηματοδότησης μέχρι την εκλογή του νέου κοινοβουλίου. Αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε άτεκτοι και έτσι λοιπόν τι πετυχαίνουμε τα μακροπρόθεσμα προγράμματα για την ανάπτυξη της υπέτρου να μπορούν να συνεχιστούν. Και εδώ από πλευρά αβεβαιότητας και ανασφάλειας ε, στα πλαίσια του πολιτού νομιστομικού πλαισίου δεν υπάρχει συμφωνία για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Στις τεχνικές συζητήσεις ε, έχουμε μια διατύπωση, ψάχνουμε μια διατύπωση για μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το λέω ξεκάθαρα, δεν μου φτάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γράφει σε τέτοιε δηλώσει ότι σκοπεύουμε να κάνουμε το χύψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επιφανειακό. Έχουμε όλε τις καλές προθέσεις του κόσμου σε πολλά θέματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη πώς να το κάνουμε σε ό,τι αφορά την οριζόντια κανονισμό προχωρήσαμε καλά, σε ό,τι αφορά την υποστηρίξη των αποθυμάτων του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πολιτική δήλωση σε ό,τι αφορά το μηχανισμό χρηματοοικονομική πειθαρχία τη επόμενη ε, μεταρρύθμιση να βελτιωθεί το αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, κοινή αγορά. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ο κ. Νταντά μας ε, βοήθησε στα πλαίσια των τεχνικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρούμε κοινέ θέσει οι οποίε εγκριθήκαν από μεγάλη πλειοψηφία για να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα λειτουργεί για την ενέσχυση των ε, ε, αγροτών που προωθούν την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική η αλυσίδα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή για να υπάρχει και ισορροπία μεταξύ του παραγωγού και του μεταποιητή και του εμπορίου τροφίμων από την άλλη και να αρθούν τα εμπόδια. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να προβούμε σε αντίληψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Η Επιτροπή το πρώτο ήμιση του 2018 δεσμεύεται να κάνει πρόταση προς το Κοινοβούλιο. Αλλά έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να προωθήσει το θέμα αυτό, αν θέλουμε πραγματικά να πετύχει κάτι. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έπρεπε να έχουμε προτάσει. Θεωρητικά έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο αυτό, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εξακολουθούν να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυσκολεύουν τα πράγματα. Έχουν προβλήματα. Η Γενική Διεύθυνση φαίνεται ότι δεν συμφωνεί, αλλά πιστεύω ότι διαβάζοντας τις συνθήκες ε, ο τομέα αρμοδιότητα είναι κυρίω στο αγροτικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν ίσω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον πρόεδρο Γιούγκερ. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια ρύθμιση που θα βοηθήσει τους παραγωγούς, τους μεταποιητές και τις ενώσεις. Ευχαριστώ την ομάδα για την καλή συνεργασία, το επικοδομητικό πνεύμα και ο κ. Τεντά, η κυρία Μούλερ από όλες τις ομάδες συνεργασία είναι καλή και νομίζω ότι είναι καλή πρώτος, επόμενος τρομερής διάλογος. Ε, ελπίζουμε να είναι και ο τελευταίος. Αλλά δεν είμαι και πολύ βεβαίως, Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο αν δεν δείξει διάταση και πρόταση συνεργασία και διαπραγμάτευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ φοβάμαι θα υπάρχει και άλλο τριμερή διάλογο. Έχουμε επαρκή χρόνο διαπραγματευτούμε αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ δυναμική η εντολή μα από πλευρά τη Επιτροπή Γεωργία. Αποφασίστηκε αυτό με μεγάλη πλειοψηφία, το ίδιο και από όλο το Κοινοβούλιο. Ω ομάδα λοιπόν θα είμαστε πολύ σκληροί στι διαπραγματεύσει μα. Δεν θα επιτρέψουμε να υπονομευθεί το Κοινοβούλιο. Θα βρούμε καλές λύσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν τους γεωργού μα στην Ευρώπη. Είναι κατεπηγόντω λοιπόν απαραίτητο να γίνουν οι συγκεκριμένε αλλαγέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη ο συνάδελφο Άλμπερτ ε, ε, ε, ενημέρωσε την Επιτροπή, είπε αυτά που έπρεπε να πούνε. Εγώ θα ήθελα μονάχα να υπογραμμίσω ότι έγιναν πολλά σημαντικά βήματα προς τα εμπρός και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, DG Agri για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα και ευελπιστώ, ελπίζω τα τελευταία σημεία τα οποία παραμένουν σε εκκριμότητα να μπορέσουν στον τελευταίο τριμερή διάλογο να υπερκε την επόμενη Πέμπτη 12 του μηνός, όπως είπε και ο Σλάβος Ντες. Ευελπιστώ ότι αυτή η άσκηση ε, θα υποστηριχθεί και από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, γιατί το τρίτο κεφάλαιο του Omnibus ε, αναφέρεται ακριβώς στις προτάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διότι είναι συγκλίνουσες οι απόψεις αυτές και επομένως ειλικρινά ευελπιστώ να μην υπάρξουν περαιτέρω αναβολές. Εμείς πάντως σε κάθε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι και για τις διαπραγματεύσεις, για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, εις περίπτωση κατά την οποία ε, δεν ε, ε, εφαρμοστεί πλήρως η πρόταση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην τελική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σένερα. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα προς το τέλος της ε, ενημέρωσης του κυρίου Ντέσιμου στην Επιτροπή Αλίας και δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Έχω μία ερώτηση για την τροπολογία 2 που μιλάει για την υπεροχή των ε, στόχων της ΚΑΠ έναντι των κανόνων ανταγωνισμού. Συζητήθηκε αυτό το σημείο. Διατηρείται πώς έχουν τα πράγματα. Ε, θα θέλαμε να στηρίξουμε και να παραμείνουμε στην τροπολογία αυτή, γιατί είναι πολύ σημαντική. Μην την εγκαταλείψετε, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 69, που αφορά την αναγνώριση των βοσκοτόπιων. Θέλουμε οι ζώνες με βοσκοτόπια να μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις της ΚΑΠ. Πώς πάνε συζητήσεις για το θέμα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσουμε την έννοια του ενεργού γεωργού. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πρωταρχικό μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να εδράζεται η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Επίσης, ποια είναι η θέση μας ε, ως προς το σημείο που θα σας πω, γιατί δεν θέλουμε δημόσια κονδύλια να στηρίζουν ιδιωτικά προγράμματα ασφαλίσεων που θα εξασφαλίζουν εισόδημα. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ προτάσεις. Θέλουμε προτάσεις που θα στηρίζονται σε ενεργές πολιτικές που θα διασφαλίζουν το γεωργικό εισόδημα. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Οπότε κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ, εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία έχει το λόγο. Ευχαριστώ και καλησπέρα σα. Θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια για τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε ο κύριος Δες, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο και στους προηγούμενους τριμερείς διαλόγους και στις τεχνικές συναντήσεις και διευθετήσαμε πολλές εκκρεμότητες. Όπως γνωρίζετε και εσείς και οι και κύριε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε λίγο χρόνο για να αποκρισταλώσει τη θέση της ως προς τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αφορούσαν την αρχική μας πρόταση. Δηλαδή για το πρασίνισμα, τους κανόνες ανταγωνισμού και κανένα δυο άλλα θέματα. Τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη βάση για επικοδομητική συνεργασία στον επόμενο ε, τριμερή διάλογο την Πέμπτη που ευελπιστώ ότι θα είναι και ο τελευταίος γιατί όλα είναι επιτάπητος, τα συζητήσαμε εκτενέστατα, θεωρώ ότι έχουν οριμάσει τα πράγματα ώστε να καταλήξουν και τα τρία θεσμικά όργανα σε ε, μια καλή συμβαστική λύση για το σύνολο του πακέτου του Omnibus. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, φυσικά δεν είμαστε απομονωμένοι. Ε, έχουμε ένα τμήμα του πακέτου και θέλουμε το ευρύτερο πακέτο να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Οπότε είναι προς το συμφέρον μας εμείς να διεκπαιρεώσουμε το δικό μας τμήμα ώστε να βάλουμε το λιθαράκι μας σε αυτή την ευρύτερη διαδικασία. Πάντως για όλα τα σημεία που ανέφερε ο κύριος Ντες, ε, παράταση των προγραμμάτων για την ανάπτυξη πέθρου, το θέμα του αποθεματικού κρίσης, όλα αυτά τα εξετάσαμε ενδελεχέστερα και υπήρχε μια αμυδρή πρόθεση που δεν είναι αρκετή για τον κύριο Ντέσο ως προς την παράταση των προγραμμάτων για την ανάπτυξη πέθρου. Το σημειώσαμε και έχω, εκπονούμε ένα κείμενο για τη δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ευελπιστώ ότι θα διαθετηθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητε που απέμειναν στον επόμενο τριμερή διάλογο που ελπίζω να είναι και ο τελευταίος. Σας ευχαριστούμε θερμά και τώρα ο κύριος Ντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω κι εγώ με τον κύριο Νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοτομητική συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί κάτι καινούργιο από διαδικαστική άποψη. Αν υπάρχει προθυμία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα προσεγγίσει σε κάποια ζητήματα, ασφαλώ και μπορούμε να τελειώσουμε στην επόμενη τρομερή διάλογο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή. Γεωργίας θα είμαστε πιο γρήγοροι σε ό,τι αφορά την εργασία μας από την Επιτροπή Προπολογισμού και σίγουρα δεν θα είμαστε αυτοί που θα καθυστερήσουμε την όλη διαδικασία σε ό,τι αφορά την ερώτηση της ε, κυρίας Σέντρα. Κάτι δεν κατάλαβα σωστά σε ό,τι αφορά τις ε, εκτάσει αυτέ, αλλά κοιτάξτε τα πράγματα διαφέρουν πολύ από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Στη Γερμανία λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν ε, ασφάλειες ε, ανασυνεταιρισμό η οποία οι οποίε σκοπό έχουν την ελεγχιστοποίηση του κινδύνου και θα πρέπει ασφαλώς να αναμένουμε την ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων σε κράτη-μέλη αλλά υπάρχει σαφής απόφαση του Κοινοβουλίου την οποία και ακολουθεί πιστά η διπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κατά πόσον θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι, κάποιο στοιχείο επιπλέον, αλλά κατά τα άλλα ισχύει η εντολή στην διαπραγματευτική ομάδα. Και κύριε Σονέρα, αν θέλετε να μου εξηγήσετε αυτό που είπατε για τις ε, χερσαίε εκτάσει. Ευχαριστώ. Μπορεί και απευθείας να σας εξηγήσει η κυρία Σένερα ε, τι ε, ρώτησε και τι εννοούσε. Μπορείτε διμερώς να τα ξεκαθαρίσετε. Ε, εξαντλήσαμε την απογευματινή μας σε διάταξη. Αύριο το πρωί θα έχουμε τις ψηφοφορίες, οπότε μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίες. Ε, θα ξεκινήσουμε στις 9 και μετά την ε, ψηφοφορία θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Ευχαριστώ τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους όσοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ.